Good afternoon everybody. Um, Καλησπέρα. Είναι 3 και 10. Ε, θα περάσω στα σουηδικά. Αν θέλετε να με ακούσετε και να με καταλάβετε, μπορείτε να να κρατήσετε, να αλλάξετε, να βάλετε ακουστικά. Όσοι καταλαβαίνετε σουηδικά δεν χρειάζεται. Οι υπόλοιποι αλλάξτε παρακαλώ. Καλώς ήρθατε. Θα ξεκινήσουμε το σημείο 1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν έχουμε λάβει προτάσεις για τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης. Προτείνω λοιπόν να την υιοθετήσουμε. Σημείο 2. Ανακοινώσει του Προέδρου. Θα βρείτε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης ε, των συντονιστών στους φακέλους σας. Και αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρούμε ότι αυτά τα πρακτικά είναι υιοθετημένα. Αύριο 21 Ιουνίου θέλω να σας θυμίσω ότι η Επιτροπή θα ξεκινήσει μια εκστρατεία διετή που αφορά τις γυναίκες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Ο στόχος είναι να συμμετάσχουν περισσότερες γυναίκες στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Και τα μέλη βεβαίως της Επιτροπής μας είναι πρόσδεκτα στις 9.30 αύριο λοιπόν θα γίνεται εγγένεια αυτής της ε, εκδήλωση, αυτή τη εκστρατείας, τη διετούς εκστρατείας της Κομισιόν. Τελευταία ανακοίνωση. Το Προεδρείο αποφάσισε να καταστήσει την διερμηνία πιο αποτελεσματική, μάλλον να τη χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικά, για να το πω έτσι. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να συνεδριάζουμε από εδώ και πέρα μόνο Δευτέρα και Τρίτη. Μόνο Δευτέρα και Τρίτη μπορούμε να έχουμε διερμηνία στις γλώσσες που επιθυμούμε. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον θα πρέπει να ψηφίζουμε Τρίτη πρωί, από τις 9 η ώρα. Κάτι τη διάρκεια βέβαια της εβδομάδας των Επιτροπών, εννοείται. Περνούμε τώρα στα επόμενα σημεία της σημερινής διάταξης. Βλέπω ότι η κυρία Παπαδοπούλου έχει φτάσει καλώς ήρθατε. Θα συζητήσουμε την θέσπιση του προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία και την γνωμοδότησή της, βεβαίως. Και θα της δώσω αμέσως το λόγο. Κυρία Παπαδοπούλη, έχει το λόγο. Μικρόφωνο, Μικρόφωνο παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Είχα μια πολύ σημαντική συζήτηση με τους κοιόδης εισηγητές για το Ευρωπαϊκό Έτος Ιθαγένειας και τη σχετική έκθεση. Ε, μόλις τελειώσαμε το διάλογο που δεν ήταν εύκολος. Τώρα το σημερινό μας θέμα είναι η δημιουργία του Ορίζοντα 2020 που είναι το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία από το 1914 μέχρι το 2014 μέχρι το 2020. Το πρόγραμμα αυτό θέλει να εξασφαλίσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης είναι το χρηματοδοτικό μέσο για την εφαρμογή της Ένωσης της Καινοτομίας, που είναι ε, μία από τις 7 εμβληματικές ε, πρωτοβουλίες της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Από το 2014 2020 ε, θα έχουμε 8 δισεκατομμύρια ευρώ στη διάθεσή μας και το Horizon 2020 θέλει να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη στην Ευρώπη μέσω της αριστείας στην έρευνα και στην καινοτομία. Θέλουμε να ενισχύσουμε τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ για την έρευνα και την κοινοτομία, κάτι που είναι πολύ φιλόδοξο και είναι σημαντικό. Η προώθηση τη ισότητα των φύλων στα πλαίσια αυτά. Και η διάσταση του φύλου επίση να ληφθεί υπόψη. Μέχρι το 2020 θα χρειαστούμε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο περισσότερου ερευνητέ. Για να επιτύχουμε το στόχο, οι προποθέσει του νέου προγράμματο θα πρέπει ε, να μην ε, είναι, έχουν προκατάληψη εναντίον κάποιου φίλου. Θα πρέπει να γίνουν ε, πολλές προσπάθειες, ούτως ώστε να ανοίξει το πρόγραμμα σε περισσότερους συμμετέχοντες και κυρίως σε, περισσότερες, σε περισσότερες επιστήμονες, γυναίκες δηλαδή, από όλη την Ευρώπη. Για να εξασφαλίσουμε λοιπόν αυτή την επιστημονική αριστεία και την τεχνολογική καινοτομία, σε αυτή την προσπάθεια για την έρευνα στο μέλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξήσει ουσιαστικά τον αριθμό των ερευνητών, ερευνητριών δηλαδή, γυναικών, μέσα σε αυτό το ένα εκατομμύριο επιπλέον ερευνητών που χρειαζόμαστε. Στη τροπολογίες μου κυρίως ε, μιλάω ε, για την διάσταση του φύλου στον ορίζοντα 2020, ούτω ώστε να δώσουμε ίσε ευκαιρίες και στα δύο φύλλα, στον τομέα της έρευνα, να εκπροσωπούνται δηλαδή στην έρευνα, στην ε, κινητικότητα και να έχουν επαρκή κονδύλια. Στην έκθεσή μου επίσης λέω ότι το θέμα του φίλου θα πρέπει να είναι παρόν στις τρεις προτεραιότητες του 2020 για την αριστεία, για την, τον ηγετικό ρόλο στην ε, βιομηχανία και στις προκλήσεις της κοινωνίας. Θα πρέπει επίση να απεικονίζετε στην κατανομή τη χρηματοδότηση μέσω ε, των δικτών για, τους, ε, για τα φύλλα, ούτω ώστε να εκπροσωποιούνται ε, στην έρευνα πιο ισορροπημένα ισορροπημένα γυναίκες. Η περισσότερη χρηματοδότηση στον τομέα τη Έρευνα πηγαίνει σε άντρε και όχι σε γυναίκε. Και αυτό είναι εμπόδιο το οποίο θα πρέπει να καταπολεμήσουμε. Υπάρχει και ένα άλλο εμπόδιο, τα ανώτατα όρια. Έχουμε πολλές ε, γυναίκες που έχουν πολύ ταλέντο, ε, είναι καλές επιστήμονες, έχουν πάρα πολλά προσόντα, αλλά δεν προάγονται όμως. Ε, γιατί τελικά τις παίρνουν οι άντρες, οι αδελφοί τους. Αυτό είναι ένα τεράστιο εμπόδιο, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουν, αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με φιλοδοξίες και εμείς θα πρέπει επίσης να το καταπολεμήσουμε. Υπάρχει υπεκπροσώπηση των ε, ερευνητριών σε ηγετικέ θέσεις ε, στον τομέα της έρευνας και της ε, καινοτομίας και αυτό το φαινόμενο είναι πολύ διαδεδομένο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα, σε, ερευνητικά προγράμματα και σε επιστημονικούς τομείς, όχι μόνο σε συμβουλευτικές ομάδες, αλλά σε όλες τις δομές ε, που υπάρχουν στα πλαίσια του ορίζοντα 2020. Το EITRC, το JRC, οι κατευθύνσεις ομάδες, οι ομάδες υψηλού επίπεδου, οι ομάδες εμπειρογνωμόνων και τα λοιπά. Σε τα πανεπιστήμια, στα ερευνητικά κέντρα, στα ερευνητικά ιδρύματα, γιατί και εκεί βλέπουμε ότι κυριαρχούν οι άντρες. Δεν βλέπουμε πολλές γυναίκες παρούσες. Επίσης, δεν θέλουμε ε, να υπάρχουν τομείς έρευνας για άντρε και άλλοι για, για γυναίκες. Στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα θα πρέπει να προωθήσουμε την ιδέα ότι η επιστήμη ε, αφορά και τα δύο φύλλα. Και τα δύο φύλλα πρέπει να δραστηριοποιούνται, όχι μόνο οι άντρε. Και τέλος, λαμβάνουμε υπόψη το ότι, φάει, ότι υπάρχει μικρό ποσοστό ε, εκπροσώπηση των γυναικών ε, στο 5ο και 6ο πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020, ούτω ώστε να προάγονται επαγγελματικά και οι άντρε και οι γυναίκε και να έχουν τι ίδιε ευκαιρίε. Επίση, να εστιάσουμε στην κινητικότητά του και στον τρόπο που μπορούμε ε, να συμφιλιώσουμε την οικογενειακή ζωή και την επαγγελματική ζωή. Αυτέ τι ιδέε προωθούμε με τι τροπολογίε μου και περιμένω να ακούσω τι απόψει σα, ούτω ώστε να δω πώ θα γίνει καλύτερη αυτή η έκθεση και να προωθεί πιο αποτελεσματικά την ισότητα. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να στέκανε στον λόγο. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, να καλωσορίσω μια ομάδα επισκεπτών που προσκάλεσε η κυρία Λοχπίλερ. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Είναι καλό να έχουμε και κοινό στην Επιτροπή μας. Κυρία Μωράν Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομη. Απλώς να ευχαριστήσω την κυρία Παπαδοπούλου που αφοσιώθηκε τόσο πολύ στο θέμα αυτό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα πρέπει να τονίσω την σημασία αυτή, διότι τόσο τα κράτη όσο και οι οικογένειες επενδύουν ιδιαίτερο στην μόρφωση των παιδιών τους, αγοριών και κοριτσιών. Τα κορίτσια σήμερα έχουν πολύ καλή εκπαίδευση και μόρφωση. Όμως όλη αυτή η προσπάθεια αποδίδει μόνον εάν τους επιτρέπουμε να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία και μάλιστα υψηλού επίπεδου στην έρευνα δηλαδή ο προσανατολισμός των νεαρών κοριτσιών, των σπουδαστριών προς την έρευνα, πρέπει να είναι πολιτικός στόχος και νομίζω μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε πολιτικό στόχο αρκετά περιοριστικό, ε, δεσμευτικό, διότι διαπιστώνω ότι τα κράτη-μέλη απαιτούν από τον ιδιωτικό τομέα σε μεγάλο ποσοστό πράγματα που οι ίδιοι δεν τα εφαρμόζουν στη δημόσια διοίκηση. Οπότε στον τομέα της έρευνας που το γνωρίζω καλά, διότι αυτή ήταν η επαγγελματική μου σταδιοδρομία, βλέπω ότι οι άντρες κατέχουν τις κορυφαίες θέσεις στην επαγγελματική πυραμίδα, ενώ οι γυναίκες εργάζονται στον τομέα της έρευνας σε χαμηλότερα κλιμάκια και με μικρότερη προβολή στα μάτια της κοινωνίας ή υποβιβάζονται σε θέσεις μικρότερης σημασίας. Η έκθεση λοιπόν αυτή υποκρύπτει αντιγόνη την νόμιμη θέση των γυναικών στα υψηλότερα κλιμάκια της έρευνας, της επιστημονικής έρευνας, σε όλους τους ερευνητικούς τομείς. Εκτίμησα ιδιαίτερα την καταπολέμηση του, της γυάλινης οροφής, διότι εν μέρη αυτό είναι αλήθεια, οι γυναίκες έχουν την τάση να υποτιμούν τον εαυτό τους, να αμφισβητούν τον εαυτό τους για το κατά πόσον μπορούν να κατέχουν τη μία ή την άλλη θέση. Πιστεύω όμως ότι αυτό το επιχείρημα είναι εύκολο να χρησιμοποιείται για να παραμένουν οι γυναίκες παγιδευμένες σε χαμηλότερα κλιμάκια και να μην μπορούν να αναρριχηθούν στην ε, κλίμακα της σταδιοδρομίας και της ιεραρχίας. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε σε όλους τους τομείς την ευκαιρία αυτή που έχουμε με την ισότητα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ανδρών και γυναικών. Βλέπουμε ότι οι γυναίκες έχουν σταδιοδρομίες πολύ λιγότερο εξελίξιμες από ότι οι άνδρες. Και επίσης κάτι άλλο που πολύ σωστά καλύφθηκε από την συνάδελφο, την Αντιγόνη, είναι ότι δεν θα πρέπει να υπερβούμε κάποια όρια αλλά θα πρέπει να είμαστε πιεστικοί με τα κράτη και να, είμα, να δείξουμε πυγμή, διότι το όλο θέμα καθυστερεί. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Συγήτρια, η οποία μας ε, παρουσίασε τις θέσεις της. Ορίζον 2020 σε στόχο έχει να βελτιώσει το μέλλον της έρευνας και εμείς ιδιαίτερα αναφερόμαστε στην προοπτική της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι δε προτάσεις της κυρίας Συγγετρής είναι ενδιαφέρουσες. Θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε την ισότητα των ευκαιριών, επί παραδείγματι, στα προγράμματα που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σήμερα, διότι βλέπουμε ότι η συμμετοχή των γυναικών στα ερευνητικά προγράμματα είναι πολύ περιορισμένη. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να διατυπωθούν κάποιες τροπολογίες για να υπογραμμιστούν περαιτέρω αυτοί οι στόχοι. Θα πρέπει δηλαδή στο μέλλον να έχουμε πιο πολλές γυναίκες και άνδρες βέβαια στις διαδικασίες, ε, στα ερευνητικά προγράμματα, στα σχέδια για το μέλλον. Αυτό υπογραμμίζουμε εμείς με την ε, τροπολογία μας και βλέπω ότι το υπογραμμίζει και η κυρία Συγήτρη ότι δηλαδή χρειάζεται και άνδρες αλλά και γυναίκες να συμμετέχουν στην έρευνα γιατί δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι τομείς οποίους οι άνδρες έχουν υποεκπροσώπηση φερειπίν στην ιατρική σε ορισμένες χώρες. Είχα μάλιστα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε συνεδριάσεις από την Επιτροπή Βιομηχανίας μεταξύ σκιωδών εισηγητών, όπου συζητήθηκε το θέμα αυτό, το πρόβλημα αυτό. Και για τον ορίζοντα 2020 θα ετοιμαστούν αρκετές σχετικές εκθέσεις, για τις οποίες όμως αποφασίσαμε να γνωμοτήσουμε μόνο για μία από αυτές. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, ο δε ρόλος της, που μπορεί να δραματίσει η συμμετοχή, η ισότιμη συμμετοχή, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γι' αυτό θα ήθελα εγώ ως Ευρωβουλευτές να ε, αγωνιστούμε για το θέμα αυτό και ταυτόχρονα βέβαια να προσπαθήσουμε και να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και στις πολιτικές μας ομάδες, διότι εν τέλει οι πολιτικές ομάδες είναι αυτές οι οποίες λαμβάνουν την τελική απόφαση για το ρόλο των γυναικών και βέβαια τις ε, τροπολογίες που θα ε, υποστηριχθούν. Ε, θα έλεγα λοιπόν να μην περιοριστούμε μόνο στα όσα λέμε εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και περαιτέρω. Το δε 8ο ε, πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα έχει αλλάξει όνομα. Δεν είναι πλέον το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Ονομάζεται πια Horizon 2020. Η αλλαγή όμω του ονόματο δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία. Πιο μεγάλη σημασία έχει, είναι, ε, έχει η έρευνα, έχει η καινοτομία, έχει η αγορά στην οποία αποτινόμεθα και νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε. Δεν μπορούμε να μιλούμε μόνο δηλαδή για την έρευνα μέσα στο πρόγραμμα, θα πρέπει και την καινοτομία και την αγορά να υπογραμμίσουμε σαν άλλους δύο ισότιμους και σημαντικούς πυλώνες για τον ορίζοντα 2020. Okej, då undrar jag om Ευχαριστώ κυρία Willis Massich. Και ζητώ συγγνώμη για την ε, προφορά, το όνομά σας μάλλον θα το έσφαξα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πριν ε, αναφερθώ στο το 2020, ήθελα πολύ σύντομα να αναφερθώ στην, ε, στα εγγένεια της εκστρατείας στην οποία κάνετε λόγο νωρίτερα. Ε, άκουσα ότι αρχίζει στις 5, όμως όχι, στις 2.30 ξεκινάει αύριο το απόγευμα. Στο κτίριο Joseph Antal, Joseph Antal 4Q2, 2.30 το απόγευμα ξεκινάει με ομιλία της ε, κυρίας Μέρικη Κοινωνικού Επιτρόπου θα διαρκέσει δεν μια μισή ώρα περίπου η εκδήλωση. Θα μιλήσουν επίσης ο Μάρκ Ταραμπέλα από την Επιτροπή σας ο οποίος ε, θα τοποθετηθεί και θα κηρύξει και τη λήξη αυτών των εγγενείων ε, της ε, έναρξης της εκστρατείας αλλά πάντως είναι πολύ σημαντική η συνεδρίαση και ξέρουμε πως η υποστήριξη είχε λάβει και στην αντίστοιχη, στην αντίστοιχη ε, διατύπωση των προτάσεων η Επίτροπος το 2010 από την Επιτροπή σας. Επίσης μεγάλη υποστήριξη και γενικότερα για τις προτάσεις του όριζου το 2020. Για δε το πρόγραμμα πλαίσιο 7, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, προσπαθούμε εν ώψη και του το 2020 να υπογραμμίσουμε με το άρθρο 15 τη διάσταση της ισότιμης μεταχείρισης των φύλων, γιατί μέσα από αυτό το άρθρο 15 δίνουμε την, ε, υπό την ε, εστίαση στην ισότιμη μεταχείριση, στην ισότιμη συμμετοχή, όπως άλλωστε υπόθηκε και σήμερα, ανδρών και γυναικών επιστημόνων στην ε, ερευνητική προσπάθεια και την διάσταση του φύλου στην, ε, στο ερευνητικό περιεχόμενο που θέλουμε επίσης κατηδία να υπογραμμίσουμε μέσα στο ορίζοντα του 2020. Σημειώνουμε φυσικά με μεγάλη προσοχή όλα τα σχόλια που ακούστηκαν. Πιστεύω ότι είναι σύμφωνα με τους στόχους ε, που ε, επιδιώκει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτύχει με τον νόμο το 2020, ιδιαίτερα με την οριζόντια προσέγγιση, γιατί αναφέρεται και στο άρθρο 13 η ισότιμη μεταχείριση των φύλων και στις ευκαιρίες, αλλά και στο παράρτημα που ε, δίνει τα κριτήρια για όλα τα προγράμματα. Επομένως υπάρχει αυτή η αναφορά. Για δε τη λήψη των αποφάσεων και την ισότιμη εκπροσώπηση, την ισορροπημένη, όπως λέμε, ισόρροπη, όπως λέμε, εκπροσώπηση, γιατί αυτός είναι ο που χρησιμοποιούμε, σε όλες τις επιτροπές. έχουμε την ίδια προσέγγιση για δε τα ε, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα η Ινστιτούτα όταν διατυπώνει προγράμματα, ε, μάλλον έργα μέσα σε ένα πρόγραμμα όπως το πρόγραμμα πλαίσιο πλαίσιο 7 ή ορίζον 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επιτροπέ, απευθύνεται σε επιτροπέ. Και βέβαια μπορούμε να δούμε τη σύνθεση μια επιτροπή, αλλά δεν μπορούμε να επιλέξουμε εμεί απευθεία από τα ε, ερευνητικά κέντρα ή τα πανεπιστήμια. Γι' αυτό χρειάζονται τα μέσα, αυτά τα εργαλεία, τα οποία αναπτύσσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την άλλη, υπάρχει ειδική χρηματοδότηση για την χρηματοδότηση της ισότιμης ε, ε, μεταχείρισης των φύλων υπό τον ε, τίτλο κάπως συγκεκριμένη θα έλεγα καινοτομία στην επιστήμη όπου πάλι και στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο χρηματοδοτούμε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια εφόσον θεσπίζουν, ιδρύουν και υλοποιούν σχέδια, έργα, απτά για την ε, ισότιμη πρόσβαση των ε, δύο φύλων. Άρα τα χρηματοδοτούμε έτσι έμεσα τρόπον τεινά από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με διορθώσατε. Ε, δεν ήθελα να πω ότι ξεκινάει στις 5, ε, ήθελα να πω ότι τελειώνει στις 5. Ε, αλλά όντως τελικά αρχίζει 2,5. Αυτό είναι το βασικό. Άλλος, κανείς θέλει το λόγο. Όχι, τελευταία κύριε Παπαδοπούλου για να συνοψίσει. thank... Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλια τους. Ε, ευχαριστώ την κυρία Γκροστέτ για αυτά που είπε και για την κυρία Γιώχανσον ε, μίλησαν για τη γυάλινη οροφή που δεν θα πρέπει να είναι άλοθη για να μην προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των ερευνητριών γιατί χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες ε, και στον στρατηγικό προγραμματισμό και όπως είπε και ο κύριος Γιώχανσον όταν δημιουργούμε και φτιάχνουμε νέα καινοτόμα προγράμματα θέλουμε παρούσες και τις γυναίκες ούτως ώστε να προγραμματίσουν αυτές και να αποφασίσουν τι είδους καινοτόμα προγράμματα χρειαζόμαστε ε, που θα είναι κατάλληλα για τις ανάγκες της αγοράς. Και για να λαμβάνονται υπόψη είναι εξίσου και οι γυναίκες καταναλώτριες και οι άντρες καταναλωτές. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και η ισότητα ανδρών και γυναικών στον δομή της έρευνας είναι πολύ σημαντικό, γιατί καλές είναι οι ιδέες, ε, αλλά ακόμα καλύτερη είναι η χρηματοδότηση. Και πρέπει να βρίσκονται και οι γυναίκες εκεί που αποφασίζεται η χρηματοδότηση. Από μόνε τους δεν μπορούν να κάνουν θαύματα. Η Κομισιόν θα ξεκινήσει αύριο μια συζήτηση για αυτό το σημαντικό θέμα και καλό όλου σα, σε αυτή τη διετή εκστρατεία για τις γυναίκες στην έρευνα και στην καινοτομία που σκοπό έχει να υπάρξουν, να βρεθούν, να εκπροσωπηθούν περισσότερες γυναίκες σε αυτόν τον τομέα. Ε, αυτή η προσπάθεια θέλει να καταπολεμήσει και τα στερεότυπα. Θέλω να έρθετε όλοι σας αύριο, να, να παραστείτε σε αυτή την εκδήλωση, όπου θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, θα πάρουν το λόγο και διάφοροι ευρωβουλευτές και είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν οι φωνές όχι μόνο των γυναικών εκεί όπου λαμβάνονται στρατηγικές αποφάσεις, αλλά και των ανδρών οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα φύλου. Γιατί, όπως είπα, στο υψηλότερο επίπεδο που λαμβάνονται οι αποφάσεις βρίσκονται πολύ λίγες γυναίκες. Ελπίζουμε όμως ότι οι άντρες που είναι παρόντες εκεί ε, να έχουν τουλάχιστον τη θέληση να προωθήσουν την ισότητα ανδρών και γυναικών. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για να, αυτό, για να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις εκεί στο επίπεδο του στρατηγικού ε, σχεδιασμού ούτως ώστε να καταπολεθούν και τα εμπόδια που δεν αφήνουν τις γυναίκες να εκπροσωπηθούν παντού, να βρεθούν σε όλους τους χώρους. Ευχαριστώ. Τελείωσε η συζήτηση. Για το χρονοδιάγραμμα που προβλέπουμε, οι τροπολογίες μπορούν να κατεθούν μέχρι τις 25 Ιουνίου. θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 10 Ιουλίου και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Πολύ ωραία. Κλείσαμε αυτό το σημείο. Και η συνάδελφος θα πάρει τώρα την Προεδρία. Έχετε εσείς το λόγο, τη θέση και το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Και τώρα θα πάμε στο τέταρτο σημείο της ημερήσιας διάταξής μας για την έκθεση του κυρίου Γκούσταυσον για το ρόλο των γυναικών στην ε, πράσινη οικονομία, φιλοπεριβαλλοντική οικονομία. Θα σας δώσω το λόγο κύριε Γκούσταυσον για να παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που έλαβα όλες αυτές τις τροπολογίες καταρχήν. Σας ευχαριστώ που μου τις στείλατε. Ήδη στην πρώτη μου παρουσίαση, στην πρώτη παρουσίαση της έκθεσής μου, διαπίστωσα ότι δεν είναι προφανές να βάλουμε σε αυτή την έκθεση όλα όσα θα θέλαμε να βάλουμε, όσα θα ήθελα εγώ να βάλουμε. Χρειάστηκε να περιοριστούμε, γιατί είχαμε και περιορισμό σελίδων. Ελπίζω παρόλα αυτά να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο με όλες αυτές τις τροπολογίες νομίζω ότι αυτό είναι δυνατό. Υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες είναι θαυμάσιες, υπάρχουν κάποιες που θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω μέσω συμβαστικών τροπολογιών. Λοιπόν, για τις, ε, θα σας πω τώρα την άποψή μου για τις τροπολογίες και μετά θα σας δώσω το λόγο να σχολιάσετε κι εσείς. Υπάρχουν τρεις τροπολογίες. που λένε ότι υπάρχουν λάθη, που υποδηλώνουν ότι υπάρχουν λάθη στις διάφορες γλωσσικές ε, εκδοχές. Έχουμε την τροπολογία 15 του κ. Γιώχανσον, που προτείνει να τοποποιήσουμε τα δεδομένα αναφύλλω, τα σωρευτικά δεδομένα να θέλω. Τουλάχιστον στη δική μου γλώσσα, στα σουηδικά, αυτός ο όρος ε, υπήρχε. Τα σωρευτικά, ε, το aggregates δηλαδή. Υπάρχει και η τροπολογία 25 του κυρίου Γιώχανσον πάλι. Σας ευχαριστώ που δίνετε έτσι έμφαση στις λεπτομέρειες κύριε Γιώχανσον. Θέλω να πω ότι στο σουηδικό κείμενο λέμε ότι πρέπει να εισαγάγουμε προοπτικές για το φύλλο σε όλα τα θέματα του περιβάλλοντος, αλλά στο αγγλικό κείμενο λέμε πολιτικές ισότητας ή πολιτική ισότητας. Δηλαδή, οι όροι που χρησιμοποιούνται δεν είναι οι ίδιοι ακριβώ στα σουηδικά και στα αγγλικά. Θα πρέπει να τροποποιήσουμε λοιπόν τις διάφορες μεταφράσεις. Το τρίτο λάθος αφορά, αναφέρεται στην τροπολογία 55, και παρατηρώ αυτό το λάθος και εγώ χάρη στο, στην τροπολογία του κύριο Γιώχανσον. Ο κύριος Γιώχανσον ίσως θέλει να, να καταργηθεί η τροπολογία 55. Λέγεται στο σουδικό κείμενο ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν μεθόδους ούτως ώστε να ενθαρρύνουν τους άντρες να επιλέξουν τα διαδρομία τους. Ενώ στην αγγλική μετάφραση λέμε ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες, όχι τους άντρες. Ε, εγώ δεν είναι αυτό που ήθελα. Δεν να πούμε, να πούμε αυτό. Ακριβώς το αντίθετο ήθελα να πούμε. Είναι σαν να λέμε ότι θέλουμε περισσότερα μέτρα για να δουλεύουν περισσότερες γυναίκες στον τομέα της υγείας. Στην παράγραφο 23, τροπολογία 55, αυτό που έγραψα εγώ στα Σουηδικά δεν υπάρχει στο αγγλικό κείμενο, τουλάχιστον στο αγγλικό που μπορώ να τσεκάρω. Υπάρχουν λάθη που πρέπει να διορθωθούν και το τελευταίο λάθος είναι εντυπωσιακό. Γιατί ο όρος άντρε που υπάρχει στο σουηδικό κείμενο έγινε γυναίκες στο βρετανικό. Ε, ήταν γλωσσικά λάθη ούτως ή άλλως. Επίσης, κάποια πράγματα που δεν μου αρέσουν πολύ καλά. Η κυρία Γιανακουδάκη δύο φορές, μάλιστα, προτείνει να υπάρχει μία έδρα του Κοινοβουλίου. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με αυτή την άποψη. Και εγώ πιστεύω ότι είναι τρέλα να κάνουμε αυτά τα μπρο πισω ε, και τα ταξιδακια βρυξελλε Βρυξέλλες-Στρασβούργο. Αλλά αυτό τι σχέση έχει με αυτό το θέμα που μας απασχολεί τώρα, με το θέμα της εκθεσή μου. Νομίζω ότι είναι μια τροπολογία που δεν έχει θέση εδώ. Πρέπει να μιλήσουμε για γενικά θέματα. Ε, ισότητα ευκαιριών κτλ. Και ξαφνικά μιλάτε θα, για μία έδρα που θα πρέπει να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι περισσότερε. Λίγο περίεργο μου φαίνεται. Ναι. Ε, Γι' αυτό δεν μου αρέσει πολύ αυτή η τροπολογία. Εν συνεχεία, ο κύριο Γιώχανσον προτείνει να τροποποιήσουμε την κατεύθυνση της ε, έκθεσης και τον τίτλο της έκθεσης. Εγώ ήθελα να μιλήσουμε για την ισότητα των φύλων στην πράσινη οικονομία. Ενώ τελικά μιλάμε για το ρόλο των γυναικών στην πράσινη οικονομία. Άρα, επί της ουσίας μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας, αλλά τελικά πρέπει να, ίσως πρέπει να συμφωνήσουμε ότι θα πούμε ισότητα των φύλων. Τελικά όμως έχει και πολύ μεγάλη σημασία το πώς θα ονομάσουμε αυτή την έκθεση. Αν θέλετε όμως εσείς όλοι, η Επιτροπή μας, να τροποποιήσουμε τον τίτλο, τότε αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι κάπου ξεφεύγει ο τίτλος της έκθεσης. Και δεν αποφασίζουμε εμείς για τον τίτλο της έκθεσής μας, αλλά η διάσκεψη των Προέδρων. Α, των Προέδρων των Επιτροπών θα παίρνει την απόφαση, γιατί θα πρέπει να δώσει την έγκρισή της στην αλλαγή του τίτλου. Κάτι που θα μας οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Και θα ήταν κρίμα να καθυστερήσουμε για αυτό το θέμα. Και αυτό επίσης σημαίνει ότι δεν θα κλείσουμε αυτό το φάκελο τον Νοέμβριο όπως είχαμε πει και επιθυμούσαμε. Εγώ θέλω η έκθεση να είναι ώστε να τον πιο σύντομα έτοιμη. Αν το σκεφτώ το θέμα καθαρά εγωιστικά και αν μπω στη θέση της Επιτροπής, ε, σκεφτείτε ότι έχουμε μόνο έξι εκθέσεις πρωτοβουλίας. Αν ζητήσουμε τροποποίηση του τίτλου και αν διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών πρέπει να αποφασίσει, τότε όλη η διαδικασία θα μπλοκαριστεί για τις άλλες εκθέσεις και επομένως δεν θα μπορέσουμε να προετοιμάσουμε άλλες εκθέσεις πρωτοβουλίας. Αυτό το θέμα το συζήτησα με τους συντονιστές, θα πρέπει να δούμε τι άποψη έχουν οι πολιτικές ομάδες γι' αυτό. Αν αλλάξει όμως ο τίτλος, του, ο, ο τίτλος συγγνώμη, της έκθεσης, τότε θα έχουμε καθυστέρηση. Δεν θα κλείσει ο φάκελος τον Νοέμβριο, σας το λέω να το ξέρετε. Έπειτα, υπάρχουν μια σειρά από τροπολογίες που αφορούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις. Και ξέρω ότι πολλοί στην Επιτροπή μα θέλουν να, μιλούμε, να μιλήσουμε σε αυτήν την έκθεση για τι ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα ετοιμάσω μια συμβιβαστική ε, τροπολογία, ούτω ώστε να συνδέσω τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και να τι εντάξω στο υπόλοιπο, μέσα στο κείμενο, α πούμε. Ελπίζω να, δεχτείτε αυτή τη συμβιβαστική τροπολογία που θα ετοιμάσω για να ενταχθούν σωστά οι μικρομεσαίε επιχειρήσει στο κείμενό μα. Επίση, θα προσπαθήσω να συγκεράσω κάποιε τροπολογίε, όχι γιατί είναι κακέ, αλλά γιατί μιλάνε για το ίδιο πράγμα. Πολλέ τροπολογίε μιλάνε για το ίδιο πράγμα. Προσπαθήσω να τι ομαδοποιήσω. Δεν θέλω το κείμενο να γίνει πολύ μακροσκελές και πολύ περίπλοκο. Προσπαθήσω λοιπόν να τι ομαδοποιήσω. Όχι όλες, κάποιες. Τέλος. Για τι δικέ μου τροπολογίε. Αυτό... Καταρχάς, θέλω να υπάρχει σαφής ορισμός της πράσινη οικονομία είναι μια έννοια σήμερα που τη χρησιμοποιούμε όπου να είναι και σαν μαϊντανό. Γιατί ηχεί ωραία. Πάντα λέμε ότι πρέπει να έχουμε μια πράσινη προοπτική, αλλά πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας ορισμός της πράσινης αυτής της οικονομίας. Επίσης θέλω να τονίσουμε και την κοινωνική διάσταση. Όχι μόνο οικονο... οικολογική και περιβαλλοντική διάσταση, αλλά και κοινωνική διάσταση και αυτή η διάσταση πρέπει επίσης να προταθεί, προταχθεί. Η τρίτη τροπολογία που θα προτείνω. Υπάρχει στην εκθεσή μου, τέλο πάντων, λέω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τους δείκτες ανάπτυξης. Γιατί πρέπει, εκτός από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, να λάβουμε υπόψη μας Εκτός από τα οικονομικά στοιχεία και οικολογικά, περιβαλλοντικά στοιχεία κτλ. Η πρώτη τελευταία τροπολογία από τις δικές μου είναι η 61. Μιλάω για το χρόνο εργασίας. Και λέω ότι πρέπει να διερωτηθούμε αν πρέπει να παράγουμε περισσότερα αγαθά ή αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το χρόνο εργασίας που διαθέτουμε. Είναι πολύ σημαντικό να καταπολεμήσουμε και την ανεργία και τη μόλυνση. άλλα πράγματα που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας λοιπόν. Τέλος. Η τροπολογία 69. Όπου ζητάω στις αξιολογήσεις μας που κάνουμε της εξωτερικής μας πολιτικής να λαμβάνουμε υπόψη το δίκαιο εμπόριο, να λαμβάνουμε υπόψη μας την περιβαλλοντική διάσταση και τη διάσταση της ισότητας των φύλων. Νομίζω ότι αρκούν αυτά από μέρους μου και με μεγάλη χαρά θα ακούσω τα σχόλιά σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, για την πολύ σοφή αυτή παρουσίαση. Και εγώ συμφωνώ στην προσέγγιση σας ε, για τις τροπολογίες που αφορούν ε, την ε, έδρα του Κοινοβουλίου και που δεν έχουν θέση εδώ. Και δίνω το λόγο ευθύ αμέσω στον κύριο Ρωμέβα Ιρουέδα, στον συνάδελφο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μικαήλ, για την έκθεση αυτή. Θα πρέπει να πούμε ότι από τη δική μου πλευρά ήταν αρκετά απλά αυτό που είχα να κάνω. Βεβαίω διάβασα την αιτιολογική έκθεση και μετά το κείμενο, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που ούτω ή άλλω είναι θέμα κοινή λογική στη Σίγουρα κάποια σημεία μπορούν να ενδυναμωθούν, όμω είναι σημαντικό το θέμα για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί είναι ζωτική σημασία να μην ξεχνάμε την προοπτική τη ισότητα των φίλων στι πολλαπλέ τάσει που έχει η οικονομία και για την περιβαλλοντική κρίση μιλάω, αλλά και για την οικονομική και πολιτική που ζούμε. Εδώ λοιπόν υπάρχουν σαφώς αλληλοσυσχετισμοί και το έγγραφο πολύ σωστά προσπαθεί να διορθώσει τις τρεις αυτές διαστάσεις. Ε, όπως βλέπετε έχουν υποβληθεί λίγε τοπολογίε, αλλά και πάλι νομίζω ότι οι τροπολογίες αυτές και οι άλλες που, έχετε, που έχουν γίνει παραδεκτές για να βελτιώσουν το κείμενο θα οδηγήσουν σε καλό αποτέλεσμα. Δύο παρατηρήσεις. Ένα θέμα τακτικής που αναφέρατε και εσείς για τον τίτλο. Νομίζω καλό θα ήταν να γίνει αυτή η αλλαγή, γιατί και εγώ συμφωνώ. Α γίνει αυτή όμω η αλλαγή στην Ολομέλεια, για να αποφύγουμε να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Είναι τεχνικό έτσι κι το ζήτημα. Δεν ξέρω, θα μα πει και η γραμματεία. Για να αποφευχθεί αυτό ο σκόπελο που εσεί αναφέρατε. Εντάξει, μπορούμε να το συζητήσουμε και αργότερα. Και κάτι άλλο που για μένα είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ανοιχτοί ώστε να συμπεριλάβουμε και κάποια συμπεράσματα που μπορούν να προκύψουν από το Ρίο συνήκωση. Για τις πράσινες οικονομίες, σίγουρα κάποια ζητήματα θα συζητηθούν εκεί και βέβαια και στις ερχόμενες ημέρες. Πέραν αυτού, θέλω απλώς να τονίσουμε την εξής ιδέα, μάλλον δύο ιδέες. Πρώτον, το ανέφερε ο κύριος Τζόνσον όταν επέβαλε την τροπολογία του. Είναι ζωτική σημασία να καταλάβουμε ότι η κρίση έχει προκαλέσει περικοπές στους κρατικούς προπολογισμού. Είναι δραματικές οι συνθήκες της δημόσιας υπηρεσίας Σε αυτό που αποκαλούμε δημόσιες υπηρεσίες και που όπως όλοι ξέρουμε αφορούν και γυναίκες που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα. Αυτές οι δημοσιονομικές περικοπές λοιπόν που βλέπουμε να επιβάλλονται δεν αφορούν την πράσινη οικονομία αλλά την βασική οικονομία μέσων των ε, κυρίαρχων πυλώνων του κράτους πρόνοιας. Αυτός όμως ο βασικός πυλώνας του κράτους πρόνοιας δεν θα πρέπει να απειλείται όπως τώρα συμβαίνει. Και όλα αυτά αλληλοσυσχετίζονται. Είτε δούμε την περιβαλλοντική διάσταση της κρίσης, είτε όχι. Γιατί υπάρχει και η κοινωνική που συμβαδίζει. Και αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο παρελθόν. Θα πρέπει λοιπόν την διάσταση της ισότητας των φύλων να την συμπεριλάβουμε και στο πλαίσιο της κρίσης. θα πρέπει το επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας που γνωρίζουμε να διατηρηθεί. Έχετε αναφερθεί σε αυτό και το αναγνωρίζω. Επίσης κάτι άλλο σημαντικό. Προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι θα προαχθούν οι γυναίκες και ο ρόλος τους στην λεγόμενη πράσινη οικονομία, κάτι που αφορά ορισμένες φορές τομείς που, όπου κυριαρχούν οι άντρες, εκεί θα πρέπει να οργανώσουμε και τη στατική μας, ώστε ο ιδιωτικός τομέας που κυριαρχείται από τους άνδρες να ληφθεί υπόψη. Πρέπει ολόκληρη η κοινωνία να αναδιαρθρωθεί, ώστε να αποδοθεί ο σωστός ρόλος σε αυτά τα νέα οικονομικά πλαίσια Όλα αυτά τα σημαντικά σημεία ούτω ή άλλω αναφέρονται και μερικέ από τι τροπολογίες ελπίζω ότι θα τα ενδυναμώσουν στη σωστή κατεύθυνση. Δεν θα είχα κάτι να προσθέσω. Απλώς θα περιμένουμε τις συμβαστικέ προτάσεις που θα μας δώσει ο Μίκαλ και θα τα ξανασυζητήσουμε. Merci, monsieur. Σας ευχαριστώ κύριε Ρωμεύα. Μία διευκρίνηση. Ω προ την αλλαγή του τίτλου που αναφέρεται, Ξέρετε ότι ε, τον τίτλο και την έκθεση μαζί εγκρίνουμε. Άρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε στη διάρκεια της επεξεργασίας μας εκθέσεως του τίτλου ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε ολόκληρη διαδικασία για να γίνει κάτι τέτοιο. Κύριε Γιώχανσον, είχατε στήσει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Γκούσταυσορ, ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Είναι πολύ καλή. Και... Μετά τα εγκόμια προς τον εισηγητή, γιατί πράγματι είναι πολύ καλή η έκθεσή του, δεν ξέρω πώς μπορώ να διατυπώσω Πώς λοιπόν, είναι δυνατό να διατυπώσω κάποια επίκριση. Εν πάση περιπτώσει όμως έχουμε σημαντικές πρωτοβουλίες. Βιωσιμότητα οικολογική, πράσινες μεταφορές, έρευνα, τεχνολογία, εταιρική σχέση, πιο πράσινα καύσιμα. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω μπορούμε να τα καλύψουμε. Σημαντικό είναι επίσης να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο μια πιο πράσινη οικονομία θα επηρεάσει τη ζωή των ανδρών και των γυναικών σε διάφορου τομεί. Στατιστικέ λοιπόν, ανάλογα με τον τομέα, θα πρέπει να αναπτύξουμε. Και βέβαια θα πρέπει να, να χρησιμοποιηθούν και τα διαφορετικά τομεία. Όσον αφορά την ίδια την έκθεση, πρέπει να πω ότι αργά-αργά ανακαλύπτω τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν για να γίνει κάτι εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο. Εν πάση περιπτώσει ελπίζω να μπορέσει να γίνει κάποια αλλαγή στον τίτλο. Και πάντως με χαρά κύριε Σεγητή, Σεγητά βλέπω ότι συμφωνείτε επί της ουσίας στο θέμα αυτό. Φαντάζομαι και οι λοιποί συνάδελφοι της Επιτροπής μας. Εν πάση περιπτώσει ίσως το συζητήσουν οι συντονιστές στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώχανσον. Ήσασταν και σκιώδης εσύ εκ μέρους της, ε, της ομάδας των φιλελευθέρων. Κυρία Τόξεν έχει το λόγο επίσης. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και θα ήθελα να ακούσω τις ευχαριστίες μου κύριε Γκουσταυσόν για την έκθεση. Είναι πολύ σημαντική, πιστεύω. Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι ε, ιδιαίτερα θέτετε το δάκτυλο από το τύπο των ήλων για το ποιο, τι είναι το πιο σημαντικό στην υπόθεση αυτή. Θα έχουμε ασφαλώ και από τη Γενική Διεύθυνση για την Ενέργεια και από τη Γενική Διεύθυνση για το Περιβάλλον ε, να συζητήσουμε γιατί θα πρέπει όλοι θα πρέπει να τηρηθούν οι υποσχέσει που έχουν δώσει όλοι οι επιτροποί όταν, τήρησαν, όταν υπέγραψαν ε, το χάρτη για τα ε, δικαιώματα ανδρών και γυναικών ε, για τις γενικές ευθύνσεις συγκεκριμένα. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε, πρέπει να υπογραμμίσουμε αυτό που λέτε κι εσείς, ότι δεν υπάρχει υπαρκή διάσταση του φίλου στην ε, συνέχεια του Ρίου και στα μέτρα που εισάγονται εν ώψη αυτού. Και θα πρέπει να επιμείνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εισαγάγει τη διάσταση του φύλου και σχετικά τέτοια μέτρα σε κάθε πολιτική για, το πράσινο, για την πράσινη οικονομία. Γιατί πάντα μιλούμε για τα ίδια θέματα. Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώσαμε την ε, οδηγία για την αποτελεσματικότητα της χρήση ενέργεια μεταξύ Συμβουλίου Επιτροπής Κοινοβουλίου, από την οποία αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν ένα εκατομμύριο νέες θέσει εργασία, αλλά διάσταση του φύλου στις ε, θέσεις αυτές εργασία δεν έχουμε. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμήσεις για το ποιες θα είναι οι αρσενικές θέσεις εργασίας και οι θηλυκές και βεβαίως οι ουδέτερες. Για τα διαρθρωτικά ταμεία επίσης θα ήταν πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον πρέπει να αρχίσει και έχει ξεκινήσει η Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά πρέπει και εμείς να τον αναλάβουμε. Πρέπει να αρχίσει το, η προσπάθεια για την καλύτερη κατάρτιση και εκπαίδευση των γυναικών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε περισσότερη κατάρτιση για τις γυναίκες ε, στην ε, νέα περιβαλλοντική τεχνολογία και επίσης ποσοστώσεις ή άλλα μέτρα στη λήψη των αποφάσεων στα διοικητικά συμβούλια για το τομέα αυτών. Μου άρεσε πολύ η έκθεση. Merci, Madame Thompson. La parole est à Madame Η κυρία Λούλινγκ έχει το λόγο, παρακαλώ. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι δεν είμαι σκιώδη ηγετρία τη ομάδα μου. Μα και γι' αυτό δεν σα ανα... ανήγγυλα λέει η πρόεδρος ως και ηγητρία. Θα ήθελα ωστόσο να πω, μια και λείπει ο σκιοδησηγητής ή σκιοδησηγητής, δύο λόγια για την έκθεση αυτή. Για τον τίτλο καταρχάς. Άκουσα αρκετά σχόλια από τους συναδέλφους που θέλουν να γελιοποιήσουν ε, την επιτροπή μας ε, και την έκθεση και που μου είπανε κάνα τίποτα πιο γελίο δεν βρήκατε από το να κάνετε έκθεση για το ρόλο των γυναικών σε μια πράσινη οικονομία. Εν εάν μπορούσαμε τουλάχιστον στον τίτλο να αλλάξουμε και να, πούμε, να μιλήσουμε για ισότητα των φύλων. Και μια και μιλούμε για πολιτική ισότητας, Μιλάμε παγίως για ίση μεταχείριση, όχι ως προς ε, τις αμοιβές μόνο, αλλά γενικά ίση μεταχείριση ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών σε κάθε θέμα των σχέσεών τους. Επομένως, εντάξει, άμα δεν μπορούμε να αλλάξουμε κιόλας θα πρέπει να το δεχθούμε. Αλλά πρέπει πιστεύω να προσέχουμε από εδώ και και στην έκθεση και στις τροπολογίες να αποφεύγουμε αστήρικτες ε, τοποθετήσεις Φερρυπίν ότι οι γυναίκες δεν επηρεάζουν το περιβάλλον κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι άντρες les personnes les plus pauvres dans les femmes pour... Ή μετά που μας λέτε ότι στο 70% θα πληγούν περισσότερο οι γυναίκες από τις κλιματικές αλλαγές. Ε, τι είναι η τρόπο. On dit toujours qu'il y a réchauffement si les femmes pauvres. Ίσως οι φτωχές γυναίκες δεν έχουν αρκετά χρήματα για να ανάψουν τη σόμπα τους, αλλά αυτό δεν οφείλεται στο, στην κλιματική αλλαγή. Έχουμε να κάνουμε με τοποθετήσει με δηλώσεις, τις οποίες δεν αντιλαμβάνομαι. Και δεν έχουν και κανένα νόημα. Είναι μάλλον προϊόν φαντασίας. Άλλο ένα. Εκεί που λέγεται ότι υποεκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις για το περιβάλλον οι γυναίκες. Δεν ξέρω αν αυτό το έχετε πιστώσει σε κάποιες μεγάλες ε, δισκέψεις. Και στις δημοσιονομικού χαρακτήρα συζητήσεις. Ε, τι να σας πω, εάν οι δημοσιονομικές συζητήσεις ε, στόχο έχουν τη θέσπιση μια πιο πράσινη οικονομίας, φαντάζομαι ότι έχουν και τοπικό χαρακτήρα, εθνικό χαρακτήρα ή περιφερειακό χαρακτήρα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να διεκδικείτε την γνώση του ότι υποεκπροσωπούνται οι γυναίκε. Δεν είναι δυνατόν να το γνωρίζετε αυτό, όπω δεν είναι δυνατόν και σε άλλου τομεί να το γνωρίζετε. Άλλη μια δήλωση, η οποία πολύ με διασκέδασε, στη αιτιολογική σκέψη ΙΤΑ-H, εκεί όπου λέτε ότι οι γυναίκε ε, καταναλώνουν λιγότερο από ότι οι άντρε. Σε σύγκριση με του άντρε. Ε, τι να σα πω, εγώ είχα την εντύπωση ότι είναι πολύ ε, πιθανότερο το αντίστροφο και σε θέματα υγεία βεβαίω και σε άλλα. Εν πάση περιπτώσει, Ας προσέχουμε λίγο τις ε, δηλώσεις μας. Οι μου φαίνονται μάλλον αστήρικτες. Ώστε να μην επιδεινώνουμε και το γελίο, το οποίο, το, το, το, τη γελία εικόνα στην οποία έχουμε ήδη εκτεθεί λόγω και του τίτλου της εκθέσεως. Ως προς τις ε, τροπολογίες 8 ε, και 14, συμφωνώ και με τον εισηγητή και με την κυρία Ομπέμ, την Προεδρεύουσα. Ξέρετε ότι οτιδήποτε και με οδήποτε τίτλο μπορεί να δημιουργηθεί και δημιουργείται. Αυτό ισχύει για όλες τις τροπολογίες βέβαια. Γιατί μου φαίνονται αρκετά γνωστά αυτά τα πράγματα. Και τώρα βλέπουμε ότι ξαναζητάμε το ίδιο πράγμα και μιλάμε και επιπλέον για πράσινη οικονομία. Και βάζουμε πράγματα μέσα που δεν έχουν καμία σχέση με την πράσινη οικονομία. Αλλά υπενθυμίζουμε αποφάσεις, ποσοστώσεις και όλα αυτά τα οποία ήδη έχουμε χίλιες φορές πει. Όταν ο κύριος συγητής λοιπόν μας λέει ότι είναι πολλά άσχετα με το θέμα ε, τα σημεία, στο κυρίως κείμενο τη εκθέσεως, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και για τις τροπολογίες το ίδιο πράγμα. Φιλιππίνη, παριθμόν 7. όπου λέγεται ότι είναι υποβαθμισμένος και μη ανεγνωρισμένος ο ρόλος ε, της γυναίκας στην πράσινη οικονομία. Δεν ξέρω να σας πω. Εμένα στην πατρίδα μου τουλάχιστον, στην γενέτηρά μου, είναι μάλλον οι γυναίκες που ασχολούνται με την πράσινη οικονομία. Και ότι ε, είναι θύματα διακρίσεων ως προς την κοινωνική ασφάλιση, την ιατροφαρμακευτική περίθελψη, την κατάλληλη πρόνοια κτλ. Τι είναι αυτά τώρα, πού τα βρήκατε. Πάλι αστηρίκτες δηλώσεις. Κοινωνικο-οικονομικό καθεστώς χαμηλότερο από αυτόν των ανδρών οδηγεί τη γυναίκα, την εκθέτει τη γυναίκα στη βία. Τι σχέση έχει η βία με την πράσινη οικονομία. Δεν να σας πω, ίσως να φταίω εγώ που δεν έχω αρκετή φαντασία για να αντιληφθώ αυτά που έχετε, έχουν περιληφθεί στο κείμενο, τι να πω, στις τροπολογίες. Εν πάση περιπτώσει νομίζω θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην τροπολογία 19, όπου ζητείται μια διεθνής ε, συμφωνία για έναν κοινό ορισμό της πράσινης οικονομίας κτλ. Από ποιον ζητάτε αυτή την ε, διεθνή συμφωνία ή μεταξύ τίνων κρατών πρέπει να συναυθεί αυτή. Κύριε Σίγητη, θέλω να απαντήσετε τώρα στις διάφορες ερωτήσεις που σας τέθηκαν. Eh, eh, Ευχαριστώ. να αντιδράσω στις ε, παρατηρήσεις κυρίας Λούλινγκ. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας και σε όλα τα σχόλιά σας, κυρία Λούλινγκ. Υπάρχουν όμως επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι οι γυναίκες δεν επηρεάζουν τόσο πολύ την κλιματική αλλαγή όσο οι άντρες. Για, λόγω των μοντέλων κατανάλωσης ε, που είναι διαφορετικοί ειδικά μεταξύ των φίλων. Α πούμε, οι άντρε χρησιμοποιούν περισσότερο το αυτοκίνητο. Κινούνται πολύ περισσότερο με το αυτοκίνητο από τι γυναίκε. Γιατί το είδο κατανάλωση των ανδρών και γυναικών δεν είναι το ίδιο. Ε, καταναλώνουν περισσότερο ενεργοβόρα προϊόντα οι άντρε από τι γυναίκε. Ε, αυτά είναι επιστημονικά δεδομένα, είναι στοιχεία που υπάρχουν δεν τα λέω εγώ. Σε ό,τι αφορά το θέμα της κλιματικής αλλαγής, φυσικά είναι ένα επιστημονικό θέμα που δεν έχει φύλλο. Αλλά οι συνέπειες του ε, είναι διαφορετικές, ανάλογα με το αν έχουμε να κάνουμε με άντρες ή με γυναίκες. Όταν χάνεται η ύπεθρος, όταν εμφανίζονται ασθένειες, αυτε αυτές είναι επιπτώσεις, είναι παρεμπίπτοντα πράγματα επιπτώσεις μάλλον του, της κλιματικής αλλαγής και οι ε, μελέτες δείχνουν ότι πλήττονται περισσότερο οι γυναίκες από τους άντρες. Καταρχάς το 70% των φτωχών αυτού του πλανήτη είναι γυναίκες και επομένως οι γυναίκες θίγονται περισσότερο από αυτές τις αλλαγές ακριβώς γιατί είναι μεταξύ των φτωχότερων αυτού του κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο λέω ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν φύλλο παρότι το, θέμα της κλιματικής αλλαγής από μόνο του δεν έχει φύλλο. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι οι άντρες ε, καταναλώνουν περισσότερο, καταναλώνουν πιο ενεργοβόρα προϊόντα κτλ. Φυσικά δεν είναι όλα άσπρα ή μαύρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι άντρε που είναι και πλούσιοι φταίνε για τι εκπομπέ του διοξιδίου του άνθρακα και οι γυναίκε είναι μονίμω τα θύματα. Δεν είναι σωστό αυτό, είναι μανιχαϊστικό, αλλά υπάρχουν κάποια επιστημονικά δεδομένα σε ό,τι αφορά την υποεκπροσώπηση των γυναικών στις αποφάσεις για το περιβάλλον και για τα δημοσιονομικά θέματα. Είναι προφανές ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται. Μετρήστε τους άντρες που είναι γύρω από, μια, από, από ένα τραπέζι που λαμβάνονται αποφάσεις. Και γιατί το συζητάω αυτό. Γιατί συμπεριφερόμαστε διαφορετικά και έχουμε διαφορετικές επιρροές και επηρεάζουμε διαφορετικά τους διάφορους τομείς δραστηριότητας. Έχουμε διαφορετική προσέγγιση του τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, του τι πρέπει να αλλάξει, του τι πρέπει να μείνει το ίδιο. Αν το 50% του ανθρώπινου πληθυσμού εκπροσωπείται στους χώρους λήψης των αποφάσεων, αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε καθόλου υπόψη ότι είναι σημαντικό για το υπόλοιπο μισό. Αν εκπροσωπούνται και τα δύο φύλλα στα τραπέζια των αποφάσεων, τότε λαμβάνουμε υπόψη και τι εμπειρίε και των δύο. Αυτό θα μπορούσε να είναι σημαντικό για την πολιτική μεταφορών. Α πούμε, για την πολιτική μεταφορά συνήθω οι άντρε αποφασίζουν για την κατασκευή ε, δρόμων, για του ποδηλατοδρόμου, για του υδροδρόμου κτλ. Οι άντρε αποφασίζουν. Οι άντρε αποφασίζουν πού θα φτιαχτεί αυτοκινητόδρομο και αποφασίζουν με βάση τα δικά του κριτήρια. Οι οδηγούν περισσότερο αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητά τους και τα χρησιμοποιούν περισσότερο τα αυτοκίνητά τους. Συχνά οι γυναίκες παίρνουν το ποδήλατό τους το... ή το λεωφορείο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας ότι η προσέγγιση στη ζωή είναι διαφορετική ανάλογα με το αν είμαστε άντρας ή γυναίκα. Ε, θα πρέπει αυτό να εκπροσωπείται και στην, στους χώρους λήψης των αποφάσεων. Ελπίζω και οι διερμηνείς να με παρακολουθούν, γιατί μιλάω τόσο φιλοσοφικά που ίσως ε, σας μπερδεύω. Ε, ελπίζω να μιλάω και πολύ γρήγορα επίσης και δεν μπορείτε να με παρακολουθήσετε. Ε, προσπαθούμε να τα καταφέρουμε. Και κάτι άλλο που ξέχασα να πω. Κύριε Ρωμέβα, είπατε κάτι σημαντικό. Είναι σημαντικό να ενημερώσουμε τα κείμενα, να επικαιροποιήσουμε τα κείμενα, επικαιροποιήσουμε τα κείμενα με βάση τις αποφάσεις του θα στο Ρίο και με βάση τις αποφάσεις του Ρίο συν 20. Ο κ. Γιώχανσον έφυγε για να μιλήσω για την τροποποίηση του τίτλου. Τέλος πάντων, όπως και εσάς κ. Λούλιν, κύριε Γιώχανσον, κύριε Ρωμέβα, και εμένα δεν μου αρέσει ο τίτλος. Αν μπορούσαμε να τον αλλάξουμε χωρίς να παρατείνουμε τη διαδικασία, θα ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος. Αλλά πρέπει να δούμε αν αξίζει τον κόπο. Δεν θέλω να μπλοκάρω όλες τις διαδικασίες τη επιτροπή μας για την αλλαγή αυτού του τίτλου. Δεν θα πρέπει όλες οι υπόλοιπε δηλαδή πρωτο, ε, να μπλοκαριστούν λόγω αυτή εδώ, μια και ζητάμε αλλαγή του τίτλου. Κυρία Τόμψαν kommissionen. Επίσης πρέπει να μιλήσουμε για το ρόλο της Κομισιόν, όπως λέτε και εσείς, σωστό. Ε, είναι ενοχλητικό το γεγονός ότι η Κομισιόν παρουσιάζει ένα κείμενο για το Ρίο Συν χωρίς να λαμβάνει υπόψη στην ισότητα των φύλων. Ενώ το συζητήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα αυτό. Το βρίσκω πραγματικά ενοχλητικό ε, για να μην πω απαράδεκτο που αυτό το θέμα δεν λαμβάνεται υπόψη. Ε, όταν ξαναμιλήσουμε για το Ρίο μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει θα μελετήσω μεγάλη προσοχή τι τροπολογίε σα. Λοιπόν, νομίζω ότι αρκούν αυτά μια και έφυγε και ο κύριο Γιώχανσεν. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Ευχαριστούμε για όλε τι διευκρινήσει που μα δώσατε. Πιστεύω το θέμα της αλλαγής του τίτλου θα μπορέσετε να το δείτε και στη συνάντηση των συντονιστών. Έχω πληροφορηθεί ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα, οπότε θα μπορέσετε να το καθορίσετε αυτό στην συνάντηση των συντονιστών. Τώρα να ακούσουμε την κυρία Γκαλό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Κατά πρώτον, να ευχαριστήσω την Επιτροπή Γυναικών και τον εισηγητή, τον κύριο Γκούσταυσον, για ένα θέμα που συχνά μας έχει απασχολήσει. Ένα θέμα που αφορά διαφορετικούς τομείς, οριζόντιου χαρακτήρα. Εδώ αφορά το θέμα αυτό την αρμοδιότητα πολλών επιτρόπων. Γι' αυτό προσέξαμε ιδιαίτερα στο σχόλιο της κυρίας Τόμψον και την απάντηση του κ. Γκούσταυσον. Θα τα μεταφέρω και στους υπευθύνου στις υπηρεσίες μας. Αυτό το σχέδιο έκθεσης λοιπόν συμπεριλαμβάνει όλου τους παραδοσιακούς όρους του θέματος της ισότητας. Αυτό δείχνει ότι δυστυχώς, οι δομέ της ε, ανισότητας που έχουν διαμορφωθεί στους περισσότερους τομείς και στην πράσινη οικονομία παραμένουν. Υπάρχει διακριτική μεταχείριση και στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές, στην απουσία των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη δυσκολία των γυναικών να συμπληρώσουν τον επιχωνιακό με τον επαγγελματικό βίο, καθώς και την ε, καταπίεση των γυναικών από την επαγγελματική τους ζωή. Εδώ, στη στρατηγική μας για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, που υιοθετήθηκε το 2010, προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη κάποιες από αυτές τις πτυχές. Όπως θα ξέρετε, με την στρατηγική αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι θα εφαρμόσει την αρχή της ευθυγράμμισης στα θέματα της ισότητας των δύο φύλων, του gender mainstreaming. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη διάσταση ισότητας των φύλων σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και σε όλους τους τομείς αναλόγως και στο πλαίσιο της εξέτασης των δικτών από την πλατφόρμα δράσης ε, του Πεκίνου, αποφάσισε η Δανική Προεδρία να εργαστεί στον τομέα των γυναικών και του περιβάλλοντος. Θα το γνωρίζετε. Ασχολήθηκαν κυρίως με τον ορισμό δικτών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ε, γυναίκες στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων, λόγω χάρη της διαπραγματεύσεως για τις κλιματικές αλλαγές αλλά και στις εκπαιδευτικές επιλογές, δηλαδή το ποσοστό γυναικών που σπουδάζουν στους επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους. Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικοί για να δούμε κατά πόσον υπάρχει ανισότητα στον τομέα του περιβάλλοντος. Τα συμπεράσματα στο θέμα, για το θέμα αυτό θα υιοθετηθούν αύριο στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ισότητα μεταξύ γυναικών, γυναικών και ανδρών έχει δημοσιεύσει και μια μελέτη για την ισότητα και τις κλιματικές αλλαγές που είναι ήδη διαθέσιμη. Βλέπουμε ότι όπως και το σχέδιο γνωμοδότησής σας, πολλά θέματα για την πράσινη οικονομία, όπως για τη μεταφορά και την ενέργεια πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται και στη μελέτη αυτή. Ευχαριστούμε, στη μελέτη αυτή ευχαριστούμε την ε, Επιτροπή Γυναικών που προέβλεψε το θέμα αυτό για συζήτηση και θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της έκθεσης. Σας ευχαριστούμε. Αν ο κύριος Γκούσταυσον έχει κάτι να προσθέσει για να ολοκληρώσουμε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Λούλινγκ, ο κύριος Γκούσταυσον δεν απάντησε στην ερώτησή μου που αφορά τη Διεθνή Συμφωνία. Ρώτησα μεταξύ ποιων συνήθει αυτή, αυτή η συμφωνία. Δεν απάντησε. Κυρία Γκούσταυσον. Τροπολογία 19. Κυρία Λούλινγκ, θέσατε συγκεκριμένο ερώτημα. Σε ποιο επίπεδο ρωτήσατε. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι ο μόνος διεθνής οργανισμός που νομιμοποιείται να προτείνει ένα τέτοιο ορισμό είναι βεβαίως ο ΙΕΦ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει από τον ΟΗΕ να ζητηθεί να συνάψει μια συμφωνία για το θέμα αυτό. Βεβαίω και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ετοιμάσει έναν άλλο κορισμό σε επίπεδο Συμβουλίου ή Επιτροπή, αλλά εξίσου σημαντικό είναι από την πλευρά τη Ένωση να προωθήσουμε αυτό το θέμα. Κατά την άποψή μου όμω ο ΟΗΕ θα πρέπει να παρουσιάσει ένα σύνολο ορισμών για την πράσινη οικονομία. Άλλωστε, η έννοια αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ομοίμορφο παντού. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται και με στρεβλές και με στρεβλούς τρόπους. Οπότε αυτό θα πρέπει να αλλάξει όχι μόνο για την οικολογία, αλλά για να έχουμε υπόψη μας και τη βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία, κύριε για αυτή την διευκρίνηση το χρονοδιάγραμμά μας ε, επηρεάζεται, διότι θα θέσετε το θέμα του τίτλου της έκθεσης αυτής στην συνεδρίαση των συντονιστών. Οπότε όλοι θα ενημερωθείτε για το νέο χρονοδιάγραμμα εργασίας ανάλογα με το τι απόφαση θα ληφθεί στη συνεδρίαση των συντονιστών. η συνεδρίαση των συντονιστών θα ξεκινήσει στις 5, διότι ακριβώ για αυτή την ώρα έχει προβλεφθεί. Οπότε ως προσωρινή πρόεδρος να σας παραδώσω και πάλι τώρα την Προεδρία, κύριε Κούσταξον. Ευχαριστώ. Οπότε λίγη η συνεδρίαση. Σας ευχαριστούμε που αναλάβατε την Προεδρία ως εισηγητή. Σας είμαι ευγνώμων. Ολοκληρώσαμε τη συνεδρίαση αυτή και θα συνεχίσουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών στις 5. Θα τα πούμε σε λίγο.